συμφωνήσετε με τη δική μου την πρόταση και να απορρίψετε τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Έληξε ψηφορία μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης. Το επόμενο σημείο σημερινής διάταξη είναι δήλωση της Επιτροπής τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης άκτα. Uh, dear colleagues, I want your attention for a minute. Για ένα λεπτό προσέξτε με παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, διότι η μερίσια διάταξη όπως υιοθετήθηκε δεν προβλέπει διαδικασία catch the eye κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής. Όμως, αν δεν έχετε αντίρρηση, προτείνω το εξή. Εάν οι ομιλητές στον κατάλογο ομιλητών τηρήσουν το χρόνο τους και υπάρχει χρονικό περιθώριο στο τέλος, τότε θα επιτρέψω να υπάρξει διαδικασία catch the eye. Υπάρχουν αντιρρήσεις από αυτού? Καλώς. Εξ ονόματος της Επιτροπής, ε, για πέντε λεπτά, ο Επίτροπος ο κύριος ε, Ντουιτ. Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε και πάλι την ευκαιρία και τη δυνατότητα να μιλήσω σε εσά για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις διαπραγματεύσεις ΑΚΤΑ. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω λιγάκι το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνονται οι διαπραγματεύσει. Η ΑΚΤΑ είναι μια συμφωνία που έχει σαν στόχο να διασφαλίσει θέσει απασχόληση στην αγορά εργασία. Αν θέλουμε λοιπόν να παραμείνουμε ανταγωνιστική οικονομία, πρέπει να βασιστούμε στην καινοτομία και στην αποκλειστικότητα διαφόρων μαρκών. Οπότε, πρέπει να έχουμε τα μέσα στη διάθεσή μας έτσι ώστε να προστατεύουμε τις ευρωπαϊκές μάρκες στις εξαγωγές. Αυτά είναι θέματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες, όχι μόνο γιατί πρόκειται για θέσεις απασχόλησης, αλλά πρόκειται και για την υγεία και για την ασφάλεια. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν διεθνείς προδιαγραφές που να είναι λογικές, ισορροπημένες και αποτελεσματικές. Και αυτό πάει πέρα από τις διαδικασίες στον ΠΟΕ για τα TRIPS. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε με αυτό. Τον Μάρτιο που μας πέρασε ήρθα εδώ και εξήγησα ποια είναι τα στοιχεία κλειδί για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις αυτές και δεσμεύτηκα υπέρ της διαφάνειας απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Και όπως βλέπετε από το σχέδιο κειμένου που απορρέει από τις διαπραγματεύσεις που γίνονται από τον Μάρτιο, είδατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τήρησε το λόγο της και τήρησε τις αρχές αυτές. Ποιες είναι αυτές. Πρώτον, ο στόχος της ΑΚΤΑ είναι να αντιμετωπίσει μεγάλες κλίμακας παραποίηση και ε, απομίμηση προϊόντων. Δεν πρόκειται μόνο, δεν πρόκειται δηλαδή για να ελέγχουμε τους ε, επιβάτες στα μέσα μεταφοράς, ε, να ελέγχουμε τα λάπτοπ τους κτλ. Δεν θέλουμε να οχλούμε τους καταναλωτές. Τώρα, αν έχετε άλλα επιχειρήματα, ευχαρίστως να τα ακούσω. Δεύτερον, η ΑΚΤΑ θέλει να ενισχύσει τις ε, προδιαγραφές που ισχύουν σήμερα όσον αφορά για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν τα τροποποιούμε αυτά. Θέλουμε να θέσουμε μίνιμουμ κανόνες για το πώς ε, θα προστατεύονται και τα δικαιώματα των καταναλωτών στα δικαστήρια. Η Άκτα θέλει να διασφαλίσει ότι οι σχεδιαστές, ε, είτε πρόκειται για μόδα, είτε πρόκειται για αυτοκινητοβιομηχανία κτλ. θα έχουν δικαιώματα τα οποία θα προστατεύονται πλήρως όταν βρίσκουμε προϊόντα ε, απομίμησης ή παραποίησης στο εξωτερικό. Υπάρχει επίσης το κοινοτικό κεκτημένο που έχει να κάνει με οδηγίες που έχουμε ήδη εμπορικές και θέλουμε να εφαρμόζεται και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά για την προστασία των δεδομένων. Η άκτα δεν πρόκειται να τροποποιήσει καμία νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε θα με ρωτήσετε, ε, και γιατί έχουμε την άκτα. Η νομοθεσία πρέπει να είναι αποτελεσματική άπαξ και όλοι έχουμε συμφωνήσει για την νομοθετική αυτή πράξη, τότε η καινοτομία θα προχωρήσει πιο άφοβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα πρέπει να ξέρετε ότι δεν θα επηρεάσουμε με τη συμφωνία αυτή την πρόσβαση σε ασφαλή φαρμακευτικά προϊόντα. Ούτε και θα υπάρχουν οι έλεγχοι γιατί είναι αυτό πάρα πολύ ευαίσθητο, ούτε θα ισχύσει συμφωνία για τις πατέντες. Σας ε, υπόσχομαι να ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από κάθε γύρο διαπραγμάτευσης, όπως το κάναμε μέχρι τώρα, θα γίνεται και στο μέλλον. Βάσει της συμφωνίας ε, πλαίσιο έχουμε ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το σχέδιο κειμένου. Θέλω επίσης να σας ενημερώσω για τον 10ο γύρο διαπραγματεύσεων άκτα που έγιναν στην Ουάσιγκτον 16 με 20 Αυγούστου. Για τα θέματα των τελωνίων υπήρξε πρόοδος. Ακόμα δεν υπάρχει αρκετή ελαστικότητα από τα διάφορα μέρη για τα πιο ευαίσθητα ζητήματα. Επίσης έγινε πολλή δουλειά για προδιαγραφές όσον αφορά την επιβολή των διατάξεων και εκεί έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει το έργο μας. Όμως δυστυχώς τους δύο τελευταίους γύρους έγινε ξεκάθαρο ότι η συνένεση όσον αφορά τις διάφορες πλευρές της άκτα θα επιτευχθεί μόνο βάσει του χαμηλότερου κοινού παρονομαστή, βάσει των πρακτικών και των συνηθιών που ισχύουν στις διάφορες χώρες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Εξαρτάται βέβαια από την φιλοδοξία τελικά που θα έχει η πράξη αυτή το αποτέλεσμα. Υπάρχουν, όπως σας είπα, πιο ευαίσθητα ε, στοιχεία και εκεί στον τελευταίο γύρο μάλλον πίσω πήγαμε, γιατί δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν για εξέδεση ευθύνη οι διάφορες πλευρές. Το ίδιο ισχύει και για τελωνιακά μέτρα, όπου πολλές πλευρές αντιτάθηκαν και έτσι δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της κυκλοφορίας προϊόντων παραποίησης και απομίμησης. Είναι απογοητευτικά βέβαια αυτά τα αποτελέσματα, γιατί εμεί θέλουμε να καλύπτεται η πνευματική ιδιοκτησία, θέλουμε τα δικαιώματα των δημιουργών να προστατεύονται. Δυστυχώς δεν έχουμε αρκετούς κανόνες που να επιβάλλουν την προστασία των διάφορων πλευρών. Μόνο το copyright πρέπει να συμπεριληφθεί στην άκτα σύμφωνα με τι τελευταίε διαπραγματεύσει. Εμεί όμω διαφωνούμε γι' αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι δεν καλύπτονται τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Τόκιο, στα τέλη του μήνα αυτού, 24 Σεπτεμβρίου με 1 Οκτωβρίου, θα γίνει ο επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να λύσουμε τα θέματα που εκκρεμούν ακόμα. Εγώ είμαι πεπισμένο πάντως ότι είναι πολύ σημαντικό συστηματικά να φροντίζουμε για την προστασία της πνευματική ιδιοκτησία σε ολόκληρο το κόσμο και πιστεύω ότι η Άκτα μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά σε αυτό. Θέλω να πετύχουν οι διαπραγματεύσεις αυτές. Τώρα, αν στα τέλη της διαδικασίας αντιμετωπίζουμε μια συμφωνία όπου δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία ουσιαστικά ή μια συνθήκη που μιλάει για πρώτης και δεύτερης κατηγορίας ε, προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, θα σκεφτούμε πολύ τη συμμετοχή μας στη συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον ε, μοναδικό γύρο μιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Ε, πρώτος ο κύριος ε, Κασπάρη για τρία λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, το 2008 είχαμε κατάσχεση Κατοντάδων χιλιάδων αντικειμένων και πολλά από αυτά ήταν επικίνδυνα. Ε, η Κίνα και η Ινδία, αυτά είναι τα μαύρα πρόβατα. Όταν έχουμε παραποίηση αυτό προκαλεί μεγάλη ζημιά στην ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και οι αγοραστέ πλήττονται. τους χάρη έχω κατά νου τα φάρμακα. Για μένα και πάρα πολλού γονεί ε, τρέμω στην ιδέα να δώσουμε στο παιδί μα ε, ένα φάρμακο μαϊμού και τελικά να πεθάνει. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα προβλήματα πρέπει να τα λύσουμε. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η πειρατεία στα προϊόντα είναι ένα θεμελιώδες θέμα. Οφείλουμε λοιπόν να προστατεύσουμε τους καταναλωτές από επικίνδυνα προϊόντα και να παρεμποδίσουμε τις οικονομικές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις μας. Γι' αυτό και εγώ χαιρετίζω τις, ε, ε, την έναρξη των διαπραγματεύσεων κατά της πειρατείας, της απομίμησης και της παραποίησης. Γνωρίζουμε ότι αυτή η συμφωνία δεν αποτελεί την πανάκια κατά τη πυρετή. αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε μια πρώτη διεθνή συμφωνία όπου ορισμένα κράτη ε, δρομολογούν τον αγώνα, τον πόλεμο κατά τη πυρετή και εύχομαι ε, να ακολουθήσουν και πολλά άλλα. Η δική μα η πολιτική ομάδα χαιρετίζει την αγαστή συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο από τότε που καταθέσαμε το ψήφιμά μα ε, την Άνοιξη και θα που φτάσαμε μέχρι εκεί. Όμω, δυστυχώ, κατά του τελευταίου μήνε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Τώρα υπάρχουν διαπραγματεύσει και ε, συγχαίρω τους διαπραγματευτές για αυτά που πέτυχαν. Γιατί όσοι και ακόμα και αυτοί που ασκούν κριτική δεν βρίσκουν στη συμφωνία αρνητικά θέματα. Ε, το θέμα ε, των ελέγχων στα σύνορα, το θέμα αυτό έχει επιληθεί, οι free strikes και ο έλεγχο των ιδιωτικών τμήματων και αυτό έληξε το ίντερνετ, οι αγορές, πωλήσει ε, και αυτά έχουν επιληθεί. Νομίζω λοιπόν βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή να παραμείνει άκαμπτη και να εκπροσωπεί και στο μέλλον τα συμφέροντα των Ευρωπαίων. Εγώ λοιπόν ε, το, τις παραβιάσεις ε, των διπλωμάτων, των δικαιωμάτων ευρυστεχνίας. Αυτά θεωρώ ότι πρέπει να τα επερασπιστούμε. Ε, σε τελική ανάλυση θα πρέπει να προστατευθούν ε, το τυρί από το τυρόλο και η σαμπάνια όπως ακριβώς και η κοκακόλα. κολα Γι' αυτό λοιπόν καλό τις Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν το μπλοκάρισμα. Ε, Σύνοδο στη Νέα Ζηλανδία κατέδειξε πώ είναι δυνατόν να ασκηθεί κριτική αλλά και πώ να αντιμετωπιστεί και αυτή. Δεν θα λοιπόν να καλέσω την Επιτροπή να συνεχίσει να ε, αγωνίζεται για την υπογραφή τη συμφωνία. Εύχομαι λοιπόν στην Κομισιόν ε, κάθε επιτυχία στον επόμενο γύρο στην Ιαπωνία και ελπίζω μετά τι διαπραγματεύσει να έχουμε μια εκτενή ενημέρωση. Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, δική μα πολιτική ομάδα ε, με, κάθε, με τη με ηρεμία θα εξετάσει τα κείμενα και κατόπιν θα καθορίσει τη θέση της σχέση με την επικύρωση της συμφωνίας. Ε, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Για τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Επίτροπε, μόλις τώρα προσπαθήσατε να μας καθυσυχάσετε. Όμως συνεχίζω να πιστεύω ότι οι ανησυχίες που εκφράζουν μεγάλο μέρος των βουλευτών δικαίως έχουν ψωθεί. Πρέπει να πω ότι τον Μάρτιο ζητήσαμε ένα ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε κατά μεγάλη πλειοψηφία προκειμένου να τροποποιηθεί το υποδιαπραγμάτευση κείμενο. Και συζητήσαμε για να ζητήσουμε τον σεβασμό του κοινοτικού κεκτημένου, την προστασία τη παροχή ε, γενώσιμων φαρμάκων και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματική ελευθερία των ε, ε, πολιτών μα. Εδώ λοιπόν οι προτεραιότητέ μα αυτέ, όσε φορέ και να τι επαναλάβουμε και τι προωθήσουμε, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη στην, στο τελικό κείμενο που θα διαμορφωθεί, ώστε να σεβαστούμε και τον κοινοβουλευτικό διάλογο που έχει διαμορφωθεί. Έτσι λοιπόν εμεί οι βουλευτέ προσπαθούμε να προβάλλουμε τι μέρε των συμπολιτών μα Ζητούμε λοιπόν, Επίτροπε, κατά προτεραιότητα να λάβετε υπόψη ότι το κοινοβούλιο που έχετε ενώπιον σας είναι συνεργάτης και όχι κάποιος που θέλει να εμποδίσει το έργο σας. Δεν θα πρέπει μόνο το απόρριτο των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο να προστατεύει την, ε, να καθορίζει την διαμόρφωση των τελικών κειμένων. Σήμερα έχουμε στα χέρια μα τη Συμφωνία ΑΚΤΑ, αλλά θα περάσουμε και ένα σημαντικό μήνυμα μετά από τη συζήτηση και την ανάγνωση και θα πρέπει να το εξηγήσουμε και στους συμπολίτε μας ε, μετά την ψηφοφορία. Η διαφάνεια λοιπόν των συζητήσεων είναι ένα στοιχείο που εμπλουτίζει τις διαπραγματεύσεις μας και απόδειξη εμπιστοσύνη. Πέραν των δύο βασικών ε, ζητημάτων, γιατί του είδου αυτοί οι πρακτικέ είναι κάτι που πλέον γνωρίζω καλά, είναι θέματα τα οποία με οδηγούν στο εξή συμπέρασμα, ότι η πρόσβαση ιδίω στα γενναιώσιμα φάρμακα είναι κάτι που θα πρέπει να προστατευτεί ιδιαίτερω, ε, ιδίω όσο την παραγωγή και την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών. Θα ξέρω λοιπόν γιατί πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή τη συμφωνία. Θα πρέπει να βελτιωθεί βεβαίω ο νόμιμο αγώνα κατά τη παραποίηση και τη απομίμηση, αλλά Υπάρχει και η συμφωνία TRIPS που μπορεί να συμπληρώσει την ε, συμφωνία ACTA. Να γίνει λοιπόν σαφή διάκριση μεταξύ των νόμιμων φαρμάκων και των ε, παραποιημένων. Ε, Επίση, το κείμενο αυτό θα πρέπει να διασφαλίσει ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των χρηστών και των νόμιμων κατόχων σα, παραπέμπω στι διάφορε διατάξει τη συμφωνία TRIPS. Και δεν μπορώ παρά να πιστέψω ότι η Συμφωνία Άκτα θα ενδυναμώσει την ευρωπαϊκή θέση στην ε, αγορά και στα εμπορικά ζητήματα. Κύριε Επίτροπε, λοιπόν, πρώτο καθήκον για μένα είναι να εξασφαλίσω ότι θα μας οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο συνένεση η συζήτηση αυτή για το υπερασπιστούμε το συμφέρον των συμπολιτών μας. Θα πρέπει λοιπόν να λάβετε και εσεί υπόψη τι δικέ μα ε, μέρημνε, όπω ε, εκφράστηκαν κατά τι διαπραγματεύσει και εκφράζονται και σήμερα, και έτσι να μπορέσουμε και εμεί να στηρίξουμε το κείμενο όπω προέκυψε από το τέλο των διαπραγματεύσεων. Οι δημόσιε διαβουλεύσει θα πρέπει να διεξαχθούν εδώ στο Κοινοβούλιο, πρωτού οδηγηθούμε σε τελική συμφωνία, και θα πρέπει να λάβετε υπόψη και το δικό μα ψήφισμα και οποιαδήποτε άλλη άποψη εκφραστεί πριν την τελική υπογραφή τη συμφωνία ΑΚΤΑ καθ' όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, άκτα fabula. Αυτό έλεγαν κατά το παρελθόν οι προγονείς μας. Ε, βεβαίως ε, νομίζω ότι έχει λήξει πλέον ε, η, το θέατρο με αυτή την συμφωνία. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι το 64% των παραποιημένων προϊόντων προέρχονται από την Κίνα. Ε, πρέπει λοιπόν να αξιολογήσουμε την κατάσταση, να δούμε κατά πόσον, ε, εφόσον δεν υπάρχουν ε, σημαντικά πλεονεκτήματα, όπω είπε και ο κύριο Επιτροπό, κατά πόσον έχει νόημα να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία. Ο λόγο που ανησυχούμε ακόμα, οι λόγοι δεν είναι πάρα πολλοί, είναι σημαντικοί. Όσον αφορά το διαδίκτυο, Ελέγχθησαν πάρα πολλά, αξιολογούμε και εκτιμούμε αυτά που είπε η Κομισιόν, αλλά συνεχίζουμε να παγρυπνούμε. Όσον αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα, αναφέρθηκε και από άλλου συναδέλφου ότι δεν είναι δυνατόν να βρούμε ε, τη χρυσή τομή ανάμεσα στα παραπημένα φάρμακα και τα, αυτά που είναι για, γενικές, ε, για γενική χρήση. Εκείνο που πρέπει να αναζητήσουμε είναι τα ασφαλή φάρμακα. Το θέμα που τίθεται είναι κατά πόσον ε, η TRIPS μπορεί να συμπεριληφθεί τουλάχιστον στο προήμιο του κειμένου της ΑΚΤΑ. Και τέλος, όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, υπάρχει μια παράδοξη κατάσταση, διότι βλέπουμε εμπόδια εμπορικά σήματα τα οποία έχουν καταχωρηθεί και θα μπορούσαν να παραβιάσουν τις γεωγραφικές ενδείξεις, αυτά την χάνουν μεγαλύτερης προστασία από τις γεωγραφικές ενδείξεις. Και εδώ λοιπόν η TRIPS προτείνει κάποια πιο συγκεκριμένη βάση, άρα δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να, είμαστε, να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση. Ευχαριστώ. ο κύριος για 1,5 λεπτό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 που η γραπτή συμφωνία ε, για την άκτα εχθές ε, έτυχε της πλειοψηφία ε, των ψήφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να στηρίζει αυτά που είπε στο ψήφισμα του Μαρτίου και κάτι άλλο. Με τη γραπτή αυτή δήλωση συμπληρώσαμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εμείς δεν επιθυμούμε να υπάρξει υπονόμευση του κανονισμού για τα πνευματικά δικαιώματα. Το κράτος δικαίου και η δημοκρατία προβλέπουν ότι η παρέμβαση στα ατομικά δικαιώματα ακόμα και στο διαδίκτυο δεν θα πρέπει να υφίσταται. Επίσης, οι υψηλέ προδιαγραφές ε, των συνταγμάτων μας, ε, της συνθήκης ε, περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η συνθήκη της Λισαβόνας εξακολουθούν να ισχύουν. Μία συμφωνία όπως είναι η Άκτα, εκείνο το οποίο πράττει είναι μάλιστα να ενθαρρύνει τα καρτέλ. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις ΑΚΤΑ βρίσκεται στο όριο της παραβίασης των συνθήκων. Αντί λοιπόν να ε, καταργήσει αυτά τα μέτρα που επικρίνουμε εμείς, τι κάνει, απλά ε, καταλήγει σε μια ε, θολή διατύπωση. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τα πράγματα είναι όλο και πιο ασαφή. Ευτυχώς λοιπόν οι αντιδράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τώρα φαίνεται να έχουν αποτέλεσμα. Με την ΑΚΤΑ, αν η ΑΚΤΑ αυτή για να πετύχει εδώ τη συμφωνία θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Τουλάχιστον από χθε πρέπει να το έχετε καταλάβει αυτό. Εξ ονόματος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριος Καμάλ για ένα λεπτό. Thank you very much, uh, Mr. President. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Καταρχάς, να καλωσορίσω τις τρεις αρχικές σας τα τρία αρχικά σα σχόλια. Πρώτα απ' όλα ότι δεν θα παραβιαστούν δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία, ότι δεν θα υπάρξουν από, το, από την πίσω πόρτα αλλαγέ στην νομοθεσία και έπειτα την υπόσχεση τη Επιτροπή ότι θα λάβει υπόψη την άποψη των διαπραγματευτικών εταίρων. Εδώ όμω πρέπει να καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ του ψηφιακού κόσμου και του κόσμου όπω είναι στην πραγματικότητα. Όπω είπε και ο κ. Άντερσον, εκδότη ε, μεγάλου περιοδικού, είπε ότι τα φτηνά ψηφιακά προϊόντα τείνουν να έχουν όλο και χαμηλότερη τιμή. Αυτό σημαίνει ότι οι βιομηχανίε του ψηφιακού κόσμου που παραπονιούνται συνεχώ πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να στηρίζονται στα παλιά εμπορικά μοντέλα, ότι θα αλλάξουν τα πράγματα και για τα δικά του προϊόντα. Όμως και σε ένα κόσμο κατασκευή προϊόντων θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι αποτελεσματική και ως και ανταγωνιστική και ω προ το κόστο του ε, εργατικού δυναμικού. Είμαστε πάρα πολύ κανεί στο σχεδιασμό των προϊόντων και κάποιε φορέ επενδύουμε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια σε νέα προϊόντα και νέα σχέδια, τα οποία όμω στη συνέχεια παραποιούνται. Ε, τα, είμαστε πολύ καλή στο σχεδιασμό αυτοκινήτων ή στα εφή e τηλέφωνα. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε ώστε τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια που επενδύονται σε αυτά τα προϊόντα δεν πηγαίνουν χαμένα. Θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή να καταλάβει ποια είναι η διαφορά μεταξύ του κόσμου του εμπορικού και του κόσμου του ψηφιακού. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, η ε, προστασία των επιχειρήσεων αυτό είναι πολύ σημαντικό, κυρίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Εγώ όμω και πάλι ε, κάνω το εξή ερώτημα. Η πειρατεία των προϊόντων μπορεί να περιοριστεί όταν στην περίπτωση όπου κάποιε χώρε, λίγε αυτέ, καταλήξουν σε μια συμφωνία. Αυτέ οι διαπραγματεύσει, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να γίνουν σε διεθνέ επίπεδο, όπω ε, παραδείγματο χάρη στον ΠΟΕ. Αυτό λοιπόν που ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ένα νέο πλαίσιο και κύριε Επίτροπε, αυτά που είπατε στο τέλο νομίζω ότι οδηγούν προ αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Επίτροπε, γνωρίζω ότι οι διαπραγματευτέ ε, τη Επιτροπή και του Συμβουλίου γνωρίζουν πολύ καλά το δίλημα και ω διέξοδο ε, θέλουν ε, οι επιχειρήσει να έχουν το δικαίωμα κατάθεση μήνυση, θέλουν σε περίπτωση που υπάρχει λόγο να μπορούν να συλλαμβάνουν του εισαγωγεί, ίσω ακόμα και του καταναλωτέ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ε, μόνο οι μικρές ε, ποσότητες μπορούν να εξαιρούνται και κυρίως ε, τα προσωπικά αντικείμενα. Αυτά είπατε. Άρα δηλαδή εσείς θέλετε να δεσμευτείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσετε μια νομική βάση όπου μια επιχείρηση που εισάγει προϊόντα η επιχείρηση αυτή εφόσον διαπιστώνει κάποιες παραποιήσεις να μπορεί να ζητήσει την καταστροφή των άλλων άλλων προϊόντων χωρίς να ε, ζητήσει ε, την ε, γνώμη της άλλης πλευράς. Ίσως αυτό μπορεί να ισχύει για κάποια κοντέινερ, όμως για θέματα όπως είναι software και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Η Microsoft, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, αυτή τελικά θα προστατεύεται και μικρές επιχειρήσεις όχι. Πολλοί λοιπόν μίλησαν για τις διαπραγματεύσεις για την άκτα και θα πρέπει να προστατεύεται η διάδοση της τεχνολογίας μεταξύ άλλων ε, και με την προστασία των αντιγράφων. Επίσης είπατε ότι υπάρχει κάποια πρόοδος και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ε, ναι μεν δέχθηκαν να συμβαστούν, όμως όσον αφορά το ποινικό δίκαιο εξακολουθεί να υπάρχει μια παραγράφος για τις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις. Ως εκ τούτου η provider αν το ζητήσει κάποια επιχείρηση είναι αναγκασμένη να δίνουν τα στοιχεία των πελατών. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις για το SWIFT διαπιστώσαμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν γνωρίζουν την προστασία των δεδομένων όπως αυτή ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν η συμφωνία δεν πρέπει να παρεμβαίνει στο δικό μας το δίκαιο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να προστατεύονται και επίσης και η προστασία των δεδομένων των χρηστών του ίντερνετ και αυτή θα πρέπει να διασφαλίζεται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σπερώνη για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο και το Συμβούλιο για αυτή τη συζήτηση. Ακόμη και πρέπει να εκφράσω τη δυσυρά μου, διότι είναι δύσκολο να συζητήσουμε γι' αυτό χωρίς να έχουμε απαραίτητα έγγραφα στη θέση μα. Στο ίντερνετ τίποτα δεν βρήκαμε και οι υπηρεσίε του Κοινοβουλίου, στις οποίες απευθυνθήκαμε, τίποτα δεν μας έδωσαν. Μας είπαν ότι η Επιτροπή έχει διαθέσει όλα τα κείμενα. Οπότε αναγκαζόμαστε να κάνουμε γενικό λόγο σε κάθε περίπτωση πάντως είναι χρήσιμο να ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Ένα θέμα το οποίο αφορά κάθε πλευρά του σχεδιασμού προϊόντων στην Ευρώπη και την προστασία των προϊόντων μας και της βιομηχανίας μας και των εργαζομένων μας. Υπάρχουν βεβαίως αντιστάσεις σε ό,τι αφορά ιδίως την διευθέτηση των εμπορικών σημάτων και των προϊόντων που είναι κατασκευασμένα σε κάποια χώρα. In, το made in. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε αν υπάρχουν μορφές θέμη ανταγωνισμού και μορφές αθέμητο ανταγωνισμού που χρησιμοποιούν την ε, χαμηλά αμοιβόμενη εργασία εργαζομένων και οδηγούν σε παραπέση προϊόντα. Είναι λοιπόν σκόπιμο να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μορφές απαράδεκτου ανταγωνισμού προκειμένου να προστατεύσουμε αυτούς που στην Ευρώπη παράγουν, εργάζονται και χάρη στην αφοσίωση, την ευφυΐα τους και τη συμμετοχή τους, στηρίζουν την Ήπειρό μας και τις προσφέρουν αυτά που χρειάζεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, η προβλεπόμενη αυτή ε, συμφωνία υποτίθεται ότι ε, θα προωθήσει την ε, διεθνή συνεργασία και επίσης και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίσει την πειρατεία. Είναι σαφές ε, ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει διαφάνεια. Τα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν στην βελτίωση της οδηγίας περί προστασίας δεδομένων, τα μέτρα αυτά όμως δεν είναι αποτελεσματικά για να αντιμετωπιστεί η πειρατεία και η παραποίηση και υπομίμηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αξιολογήσει τις συνέπειες της συμφωνίας. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη ακόμα. Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας για μένα είναι κάτι αδιαμφισβήτητο και εξίσου σημαντική βέβαια είναι και η προστασία των ατομικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωή. Ο Πέτε Χούστινγκ τοποθετήθηκε από αυτού και είπε ενώ η πνευματική ιδιοκτησία είναι πολύ σημαντική για την κοινωνία και πρέπει να προστατεύεται, δεν θα πρέπει να είναι πάνω από τα ιδιωτικά δικαιώματα για την προστασία των δεδομένων και τη ιδιωτική ζωή Και τέλο τη παράθεση. Εμεί ε, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού κάθε είδους νομική διάταξη που υπάρχει για την επίτευξη του στόχου. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, έχω οκτώ ομιλητέ ε, για το Catch Δεν πρόκειται να πάρω κανέναν άλλον και θα είμαι εξαιρετικά αυστηρό στο χρόνο για αυτούς τους οκτώ. Ε, πρώτο, πρώτη κυρία Κόστιγκερ για ένα λεπτό. Ah, Αγαπητοί συνάδελφοι, η αποτελεσματική εφαρμογή ρυθμίσεων για τη μετώπιση τη πειρατεία και την ενίσχυση τη πνευματική οδηγίας, κάτι τέτοιο βέβαια είναι θετικό. Δυστυχώ όμω, στην κοινή γνώμη υπάρχει ανασφάλεια και άγνοια. Εγώ παίρνω συνεχώς email από ανήσυχου πολίτε που λένε ότι δεν υπάρχει διαφάνεια σε αυτέ τι διαπραγματεύσει για την άκτα και η άκτα αυτή η συμφωνία επηρεάζει σημαντικά τα δικαιώματά του. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δείξουμε ότι ε, το πρόβλημα δεν είναι η άκτα ε, υπάρχει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2009 και εξ αυτής ε, απορρέει ότι ε, θα πρέπει κυρίως να προστατεύονται τα προσωπικά και ατομικά δικαιώματα. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, με βάση αυτές όμως τις συνθήκες, να μπλοκάρεται η δυνατότητα πρόσβασης πολιτών στο διαδίκτυο. Άρα δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι η άκτα, είναι το ότι μπορεί να περικοπούν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πάρα πολλά πειρατικά προϊόντα και προϊόντα παραποίησης και απομίμησης κυκλοφορούν ε, σε διάφορες χώρες του κόσμου. Πράγμα το οποίο οδηγεί σε μεγάλη απώλεια εσόδων στους παραγωγούς των αυθεντικών ε, αντίστοιχων προϊόντων είναι κάτι που αποτελεί μεγάλη απειλή για τους καταναλωτές ε, και για την αγορά εργασίας, γιατί χάνονται έτσι πολλές θέσεις απασχόλησης. Η άκτα πρέπει να είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για να αντιμετωπίζει το φαινόμενο αυτό. Συμφωνώ πάντως με τους συναδέλφους που λένε ότι χρειάζεται διαφάνεια και ότι χρειάζεται περισσότερη εμπιστοσύνη απέναντι στη συμφωνία αυτή. Πρέπει να πετύχουμε μια καλή ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των ε, καταναλωτών και την συμφωνία αυτή. Δεν μπορεί να προστατεύονται τα δικαιώματα μόνο της μίας πλευράς. Ευχαριστώ. Η εξαίρεση για τα γενώσιμα φάρμακα δεν είναι ακόμη κατάλληλη. Υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να τα επιλύσουμε. Η διέλευση των προϊόντων, ε, η μαζική εισαγωγή. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει υποχρέωση εφαρμογής της εξαίρεσης. Όταν μιλάμε για τεχνολογικά μέσα, λόγου χάρη, όσοι προωθούν και διαδίδουν τις επιστημονικές μεθόδους για να παρακάμψουν μία εξαίρεση, μία απαγόρευση, είναι Περιπτώσει που πρέπει να καταπολεμήσουμε. Πρέπει να δούμε εδώ και ποια είναι τα οικονομικά ε, θέματα που διακυβεύονται. Διότι αν δεν υπάρξει οικονομικό συμφέρον, κανείς δεν θα επιχειρήσει να παρακάμψει την ε, τεχνολογία. Επίσης πρέπει να αποφύγουμε αντιφατικές διατάξεις, ιδίω για την προστασία τη πνευματική ιδιοκτησία. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Θέλω να προσθέσω ένα νέο στοιχείο στη συζήτηση που κάνουμε για την ΑΚΤΑ. Με συνυπογράφοντας της δήλωσης 12 έχω την τιμή να σας ενημερώσω ότι η δήλωση αυτή πέτυχε μεγάλη πλειοψηφία μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ξεπέρασε τον ελάχιστο αριθμό υπογραφών. Χαίρομαι που η δήλωση αυτή θα σας φτάσει πριν τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων για την άκτα πιστεύω ότι μπορείτε να τη θεωρήσετε σαν μια εντολή για διαπραγματεύσεις από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σα υπενθυμίζω ποια είναι τα κύρια στοιχεία. Εννοείται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει διαφάνεια. Το κείμενο να δίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και πριν φτάσουμε στην επικύρωσή του. Ζητάμε λοιπόν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας να μην εναρμονιστούν εξαιτία ε, της πράξης αυτής και η ελευθερία των πολιτών, ο ιδιωτικό τους βίος και η ιδιαιτερότητα του διαδικτύου να διατηρηθούν και να δώσετε εγγύσεις γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρέπει να διερωτηθούμε σε ποιο βαθμό οι συμφωνίες αντιμετώπιση της παραποίησης ε, ίσως είναι απλά η προστασία των μεγάλων επιχειρήσεων και όχι των απλών πολιτών. Στην περίπτωση των ε, φαρμάκων ε, βεβαίως οι συμφωνίες αυτές μπορεί να προστατεύσουν τους ανθρώπους αλλά μπορεί και να καταστρέψουν και την υγεία τους. Τα παραποιημένα προϊόντα παράγονται κυρίως στις χώρες χαμηλού κόστους ε, οι κυρώσει ε, πρέπει λοιπόν να επιβληθούν απέναντι σε χώρε που επιτρέπουν τέτοιου είδου ε, πρακτικέ. Με μεγάλη μου χαρά ακούσα την Επιτροπή να διαβεβαιώνει ότι θα αντιμετωπιστούν μόνο οι παραβιάσει μεγάλη κλίμακα και όχι οι καταναλωτέ. Βέβαια, μερικοί επιθυμούν να μπλοκάρουν την πρόσβαση των ε, καταναλωτών ε, στο ίντερνετ. Γι' αυτό λοιπόν μπορούτε να μας διαβεβαιώσετε ότι οι διατάξεις αυτές ε, θα είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Κυρία Ζεντρεζιεύσκα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαίρομαι για τη συζήτηση που γίνεται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση υπέρ τη ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ω όργανο το οποίο εκπροσωπεί του Ευρωπαίου πολίτε. Θέλω να υπογραμμίσω εδώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα στην ενημέρωση πρέπει να γίνονται διαβουλευσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα εμπορίου και για εμπορικέ πτυχέ που έχουν να κάνουν με την πνευματική διοκτησία. Στη σημερινή συζήτηση άκουσα ποιο είναι το περιεχόμενο, ελπίζω να οδηγήσει σε μια καλή πρακτική και για το μέλλον. Εδώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σας για το θέμα του απόρριτου όταν πρόκειται για τις διαπραγματεύσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό στους Ευρωπαίους πολίτες εισπράτεται πολύ αρνητικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μας ενημερώνει και περισσότερο μάλιστα ακόμα για τις προσπάθειές της και μάλιστα από την αρχή. Στη γραπτή μου ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάω για τις σχέσεις της ΑΚΤΑ με... Ένα λεπτό. Uh... Κύριε Επίτροπε, μας ε, διαβεβαιώσατε ότι αυτή η συνθήκη, συμφωνεί η Άκτα, προς το παρόν δεν θα αλλάξει τίποτα όμως ε, δεν μας δίνεται τη δυνατότητα να εκφράσουμε τις δικές μας απόψεις, να σας μεταφέρουμε τις δικές μας εντυπώσεις και να παρουσιάσουμε και τις δικές μας τις ε, νομικές γνώσεις για το κατά πόσον οι παράπλευρες απώλειες ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες της Ευρώπης δεν θα είναι πολύ σημαντικότερες από ό,τι λέτε εσείς. Πρέπει λοιπόν να ε, ε, έχουμε μία λέξη, υποτίθεται, την οποία οφείλουμε να εμπιστευόμαστε. Και αν ισχύει αυτό, γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια. Γνωρίζω ότι την ευθύνη την φέρουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Όμω ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήσυχη τη συνείδησή τη. Εγώ πιστεύω πω όχι. Δεύτερο θέμα. Το θέμα τη ονομασία προέλευση. Εγώ στι διαπραγματεύσει θα καθιστούσα σαφέ ότι στην Ευρώπη κάτι τέτοιο έχει το χαρακτήρα τη προστασία εμπορικών σημάτων. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να θίξετε στη διαπραγματεύση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δύο ακόμα μιλητές και κλείσαμε. Είναι πρώτα ο κύριος Έρενχάουζερ και τέλος ο κύριος Έγκστρομ. Κύριε Έρενχάουζερ, για ένα λεπτό. Uh, kurz drei Punkte. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω τρία θέματα. Καταρχήν, ε, συγχαίρω όσου ε, συνέταξαν τη γραπτή δήλωση για την άκτα που πέρασε αυτή. Το δεύτερο, σε αφορά στη διαφάνεια, θα θέλω να απευθύνω μια ερώτηση προ τον κύριο Επίτροπο. Κύριε Επίτροπε, εσεί ε, πώ εξηγείτε ότι εμεί ω ευρωβουλευτέ εξαρτώμεθα από μια Ευρωπαϊκή Οργάνωση Πολιτών για να πάρουμε το κείμενο. Το έχω επιτέλου το κείμενο, θα το καταθέσω και σα παρακαλώ πάρα πολύ να με διαβεβαιώσετε ότι πράγματι είναι και το πρωτότυπο του κειμένου που έχω στα χέρια μου. Ε, τρίτον, ε, ευθύνη των providers ε, και διακόπτη, διακοπή, σχόλια. Δυστυχώ εμεί δεν ακούμε. Τρίτον, λοιπόν, η ευθύνη, η αστική ευθύνη των provider. Μπορείτε εσεί να μα διαβεβαιώσετε ότι θα, δεν θα εισέλθει από την πίσω πόρτα η ευθύνη των providers. Quiet, please. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Συμφωνούμε όλοι ότι η παραποίηση είναι κάτι κακό και ότι πρέπει να καταπολεμηθεί. Αυτό είναι καλό για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους πολίτες και σημαντικό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όπως πολύ σωστά ακούσαμε. Είναι θετικό λοιπόν να προστατεύουμε τα εμπορικά σήματα και την γεωγραφική προέλευση. Πολύ καλός εδώ. Όμως αυτό που είπε ο κύριος Καμίλη ότι υπάρχει μια διαφορά εδώ πέρα ανάμεσα στην άκτα και τον ψηφιακό κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι διάφοροι πάροχοι και επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε αυτό το τομέα ανησυχούν για την συμφωνία αυτή γιατί πιστεύουν ότι μπορεί να βλάψει τις εξελίξεις στον κλάδο τους. Μπορεί να βλάψει τις επιχειρήσεις και να μην μπορέσουν να προχωρήσουν στις τεχνολογίες όπως θα γινόταν αλλιώς. Οπότε κύριε Επίτροπε, προχωρήστε, καταπολεμήστε την παραποίηση, αλλά βγάλτε απ' έξω το κεφάλαιο για το διαδίκτυο. Αυτό θα ήταν η καλύτερη λύση για όλου μα. Ευχαριστώ πολύ και τώρα και να κλείσουμε τη συζήτηση εξ ονόματο τη Επιτροπή, ε, ο επίτροπο ο κ. Ντεούτ για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές που πήραν το λόγο πριν φτάσουμε στο τέλος του παιχνιδιού για την συμφωνία αυτή. Όλα όσα είπατε θα τα λάβω υπόψη μου. Να πω κάτι για το θέμα του απορρίτου. Και να απαντήσω και σε κάποιες τεχνικής φύσεως ερωτήσεις που ετέθησαν. Μία από αυτές είχε να κάνει με τη συμφωνία τρίψη όσον αφορά τη δημόσια υγεία. Κατά πόσο ρητά θα αναφέρεται στην συμφωνία ή όχι. Ναι, αναφέρεται λέει αναγνωρίζοντας τις αρχές οι οποίες αναφέρονται στην Τόχα για τι συμφωνίες TRIPS και για τη δημόσια υγεία που εγκρίθηκαν τον Εύρη του 2001 από τον ΠΟΕ στην τέταρτη διπουργική ε, συνάντηση του ΠΟΕ. Αναφέρεται λοιπόν ρητά. Επίσης, υπήρξαν και ερωτήσει για τον ιδιωτικό βίο. Και εδώ, αν κοιτάξετε το κείμενο το οποίο σήμερα συζητάμε, λέει, κατά λέξη, ότι τίποτα στη συμφωνία αυτή δεν θα πλήξει το θέμα της πληροφόρησης βάσει διεθνών συμφωνιών ή νομοθεσία που έχει να κάνει με την προστασία του ιδιωτικού βίου. Και υπάρχει και άλλη μνήμα για το θέμα αυτό στο σχέδιο κειμένου που συζητάμε επί του παρόντος, που λέει ότι για την εφαρμογή στον ψηφιακό χώρο η κάθε πλευρά διατηρεί τις αρχές που έχουν να κάνουν με την ελευθερία έκφρασης. Άρα λοιπόν ρητά γίνεται μνήα αυτών των θεμάτων στη συμφωνία. Να πω και δύο λόγια για τα φάρμακα. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα με τα φάρμακα, όχι μόνο εξαιτία της άκτα, αλλά και επειδή επί του παρόντος Συζητάμε με την Ινδία για τα θέματα αυτά. Ξέρετε ότι έχουν έτοιμα στον ΠΟΕ όσον αφορά τα φάρμακα, συζητάμε και θα καταλήξουμε σύντομα σε συμπέρασμα πιστεύω. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και καλό. Επίτροπε, διακόπτει ο Πρόεδρος. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώνουμε αυτή τη συζήτηση, γι' αυτό παρακαλώ μην κάνετε φασαρία. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε, συνεχίστε. Θέλω επίσης να προσθέσω το γεγονός ότι τα διπλώματα αυτά τεχνίας δεν καλύπτονται από την τελειωνιακή πτυχή της άκτα. Γίνεται ρητά μνήμα στην υποχρέωση αδειοδότησης, κάτι που είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Τέλος, για το απόρριτο. Δεν έχουμε πρόβλημα για να σας δώσουμε το κείμενο, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι μια πολυμερής διαπραγμάτευση και οι άλλες πλευρές πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, να συμφωνήσουν για να δημοσιοποιηθεί κάτι. Αλλά όσον αφορά το ερώτημά σας, κατά πόσο θα έχετε τη δυνατότητα να συζητήσετε την τελική συμφωνία, θα είσαστε σε θέση πριν την υπογραφή της συμφωνίας να τη συζητήσετε. Θα φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να σας περιλάβει στις διαπραγματεύσεις και θα δείτε, και στο, θα δείτε στο ανακοινωθέν τύπου για την ΟΑΣΚΔΟΝ που λέει ότι οι πλευρές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποχαρακτηρίσουν το κείμενο πριν ε, καταλήξουμε στη συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Η ζήτηση έληξε και θα προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες της ημέρας.